Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο, 3η 6 Ιουλίου 2010, από τις 9 ως τις 13, από τις 15 ως τις 20 και 30 και από τις 21 μέχρι τις 24. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου